τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με αυτό το θέμα. Έχει γίνει κάποια δήλωση, έχει ληφθεί κάποια απόφαση για δράση σχετικά με την άσκηση πίεσης στην Ταϊβάν για να καταργηθεί η θανατική ποινή. Και πότε και πώς η υπηρεσία σκοπεύει να θίξει το θέμα της θανατικής ποινής ε, στις αρχές της Ταϊβάν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί μια βασική στάση κατά της θανατικής ποινής. Ως συνέπεια των έξι εκτελέσεων στην Ταϊβάν το 2012 στις 21 Δεκεμβρίου, η Κάθριν Άστον έκανε δήλωση στην οποία καταδικάζει τις εκτελέσεις και κάλεσε την Ταϊβάν να καταργήσει την θανατική ποινή. Αυτό ήταν εναρμονισμένο με τις προηγούμενες δηλώσεις της υπατης ε, της εκπροσώπου για τις εκτελέσεις στην Ταϊβάν το 2010 και το 2011. Επ' ευκαιρία χαιρετίζουμε το γεγονός ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εσείς κυρία Πρόεδρε εκφράσατε τις ανησυχίες σας για αυτό το θέμα. Πολλά κράτη-μέλη επίσης ε, εξέδωσαν δηλώσεις με τις οποίες καταδικάζουν τις εκτελέσεις. Οι εκτελέσεις του Δεκεμβρίου προκάλεσαν μία έντονη συζήτηση στην κοινωνία της Ταϊβάν. Συζήτηση αυτή... Στη, στη συζήτηση αυτή ηγήθηκαν ε, Ταϊβάν και επιπροσθέτως, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων μια συμβουλευτικής επιτροπής ε, προς τις ε, αρχές της Ταϊβάν, που είχε το έργο να εργαστεί κατά, ε, υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής, παρετήθηκε του έργου της. Οι αρχές της Ταϊβάν όχι μόνο επικρίθηκαν για την αποτυχία τους να συμμορφωθούν με τις ε, διατάξεις της διαδικασίας της Κλεμέντζη, αλλά έδωσε, μας δίνουν την εντύπωση ότι οπισθοχωρούν στο θέμα της εκατάργησης της θανατικής ποινής. Αυτή η πολιτική τους στάση έχει εκφαστεί και στο παρελθόν. Βέβαια, το θετικό είναι ότι οι αρχές της Ταϊβάν υποσχέθηκαν να μειώσουν το πεδίο εφαρμογή και το εύρος της θανατικής ποινής και αυτό συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις όπου η θανατική ποινή ήταν υποχρεωτική για ορισμένα αδικήματα. Επίσης, οι εφέσεις από εδώ και στο εξής θα είναι ανοιχτές. Οι πρώτες ε, περιπτώσεις μας δείχνουν ότι τα δικαστήρια σκοπεύουν να θέσουν περισσότερο αυστηρές προϋποθέσεις απόδοσης της θανατικής ποινής. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θεωρεί πως η κυβέρνηση της Ταϊβάν δεν κάνει αρκετά για την προώθηση του ζητήματος αυτού και καλούμε για την άμεση ισχύ ενός μορατόριου της εκτελέσεις. Τώρα, απαντώντας στην ερώτησή σας του για το πώς και το πότε η υπηρεσία θα θίξει το θέμα της θανατικής ποινής κατά τις ε, συνομιλίες της με τις αρχές της Ταϊβάν, να σας πω ότι τώρα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάστηκαν για το θέμα αυτό και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ταϊβάν με το που αναφέρθηκε το θέμα της, ε, του μορατόριου. Μάλιστα και εγώ και ο συνάδελφος του Κοινοβουλίου ήμασταν σε αποστολή στην ε, Ταϊβάν την ε, περίοδο του Νοεμβρίου, στα μέσα Νοεμβρίου, όταν το θέμα είχε αναφερθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ταϊβάν. Μετά τις δηλώσεις της είπα της εκπροσώπου, ο κύριος Φέρι Λαπλάνς, ο εκπρόσωπος στην ε, Ταϊπέη, επικοινώνησε με τα μέλη των αρχών της Ταϊβάν και τους ενημέρωσε για τις ε, δηλώσεις του. Επικοινώνησε με τις ε, αρμόδιες αρχές της Ταϊβάν, τόνισε το ζήτημα της θανατικής ποινής και τόνισε και την επιδείνωση της κατάστασης από το 2011 και μετά και έκανε έκκληση για μελλοντική κατάργηση. Εκτός από τις ε, δημόσιες δηλώσεις και τις ε, διαδηλώσεις έχουν γίνει και άλλες δράσεις, ιδιαίτερα εκκλήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ταϊβάν προς το κοινό. Το Ευρωπαϊκό Οικονομικό ε, Γραφείο μας στην Ταϊπέη επικοινώνησε με τα μέσα ενημέρωσης για το ζήτημα της θανατικής ποινής. Απορρίψαμε κάθε κριτική για το ότι η καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την θανατική ποινή στην Ταϊβάν θα έχει οποιασδήποτε συνέπειες με τις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή. Το δικαίωμα της ζωής είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί την τον παγκόσμιο σεβασμό του. Το, γραφείο, το, Ευρωπαϊκό Γραφείο Εμπορίου και Οικονομίας στην Ταϊπέη έχει προσθέσει και στον ιστό τοπό του μια δήλωση κατά την οποία αναφέρονται οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της θανατικής ποινής. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε τον διάλογο ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στις αρχές της Ταϊβάν. Για παράδειγμα, το 2012 έγιναν δύο διαφορετικά σεμινάρια από εμπειρογνώμονες, από εισαγγελείς, δικαστές και νομικούς με ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με το ζήτημα της θανατικής ποινής. Και αυτό θα συνεχίσει και το 2013. Τέλος, η συνεργασία με την κοινωνία της Ταϊβάν σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής είναι και αυτός ένας από τους στόχους μας και υπάρχουν χρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία συνεργάζονται με μη κυβερνητικέ οργανώσει τη Ταϊβάν που αποσκοπούν στην κατάργηση τη θανατική ποινή. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που είχα για τη δήλωση. ευχαριστώ πολύ για την λεπτομερή σα απάντηση. Δεν έχω εγώ η ίδια ερώτηση, ο κύριος Τάνοκ έχει. Είμαι πρόεδρος της ε, ομάδας φιλίας του Κοινοβουλίου για την ε, Ταϊβάν ε, και πρέπει να πω ότι δεν έχουμε στην πολιτική μου ομάδα μια συλλογική θέση όσον αφορά την θανατική ποινή. Τούτου λεχθέντος να πω ότι όταν έχουμε ε, επαχθεί και προσχεδιασμένα εγκλήματα θα πρέπει αυτοί οι εγκληματίες να ακολουθούν την σωστή ε, διαδικασία. Ε, απ' την άλλη πλευρά θεωρώ ότι ε, τις, ε, τις περιπτώσεις για τις οποίες ε, αναφέρονται για την Ταϊβάν θεωρώ ότι είναι εξοργιστικό το ότι δεν αναφέρεται ότι στην ουσία αυτά όλα έχουν συμβεί στην ενδοχώρα της Κίνας από ομάδες όπως η Φέλονγκ Τάγκ και ε, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να αφαιρεθεί το σημείο αυτό εκτός και αν υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση και εν πάση περιπτώσει ε, είναι θέμα εγκληματολογικής έρευνας. Να πω επίσης ότι η Ιαπωνία και η Ινδία και οι Ηνωμένε Πολιτείες, μεγάλες δημοκρατίες και εμπορικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ακόμα, προβλέπουν ε, τη θανατική ποινή ε, είτε εξ ολοκλήρου είτε σε ορισμένα ε, από τα ομοσπονδιακά κράτη για την περίπτωση της πολιτείας, για την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, και βεβαίως ε, η κάθε χώρα έχει δικό της κράτος ε, δικαίου και έχει δικό της δικαϊκό σύστημα και βεβαίως έχει και την δυνατότητα να διατηρήσει ή να μην διατηρήσει, να καταργήσει την θανατική ποινή η θανατική ε, ποινή ακόμα και στις ΗΠΑ ε, βλέπουμε ότι ε, εξακολουθεί να είναι δημοφιλής κατά κάποιο τρόπο βεβαίως θα πρέπει να εφαρμόζεται μονάχα σε ιδιαίτερους δεχθεί εγκλήματα. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Θα θέλαμε να μάθουμε τη θέση της ομάδας σας σχετικά με τη θανατική ποινή. Ευχαριστώ. Αυτό βρίσκεται κάτω από το θέμα των ερωτήσεων. και τις ερωτήσεις δεν προβλέπεται να έχουμε πάρα πολύ ε, μεγάλη συζήτηση. Όμως πράγματι ε, πιστεύω πως πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην ε, Ταϊβάν, διότι η πλειοψηφία των κρατών χωρών έχει στην πολιτική της ατζέντα το θέμα της άρσης του μορατόριου. έτσι ώστε Σας ευχαριστώ πολύ. Όταν θα πάμε στη Γενέβη, θα δούμε εκεί, τις, συγγνώμη, Νέα Υόρκη, διορθώνει πρόεδρος, θα στείλουμε μία αντιπροσωπεία μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και μέσα στα θέματα που θα συζητηθούν θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και έμφαση στην... για την Ταϊβάν. Θα δούμε και σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούν και τα περισσότερα κράτη-μέλη και αναλόγως θα αποφασίσουμε. Σας ευχαριστώ. Τώρα έχουμε ενημέρωση για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Και πολλέ φορέ, καθώ σχεδιάζουμε το πρόγραμμα τη ημερήσια διάταξη, δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να λάβουμε πληροφορίε για τα τρέχοντα ζητήματα στι ε, διαφορέ χώρε. Προσπαθήσαμε τώρα να έχουμε μια ενημέρωση από την ΕΕΔ για τα έκτακτα ζητήματα και πιστεύω πως ε, είναι καλή στιγμή να κοιτάξουμε την κατάσταση στο Κατάρ. Το Κατάρ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, περιοχή του Περσικού κόλπου, αλλά και παγκόσμια. Διότι είναι ένα σημαντικό κέντρο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και μαθαίνουμε πολλές πληροφορίες για τον αραβικό κόσμο μέσω αυτών των μέσων. Είναι το κέντρο... Είναι τα κεντρικά γραφεία του Al Jazeera εκεί και ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις στον αραβικό κόσμο. Επίσης και η κυβέρνηση του Κατάρ θεωρεί αυτόν ε, προοδευτική δύναμη και χώρο ελευθερίας του τύπου. Όχι μόνο για το Al αλλά και γενικότερα για άλλα δίκτυα ενημέρωσης. υπάρχει έντονη επιθυμία για ελευθερία του τύπου και αυτό έχει τονιστεί από τις αρχές του Κατάρ. Πρόσφατα υπήρξε μια δικαστική απόφαση για ισόβια κάθερξη σε έναν ποιητή, τον ε, Μοχάμεντ Αλατζάμι, μετά από μια άδικη δίκη και αυτό εμείς το θεωρούμε παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. Επίσης, στο Κατάρι υπάρχει ένα νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η διατύπωση είναι αρκετά σαφής και τη βρίσκουμε και σε άλλες χώρες Και σύμφωνα με την ε, διατύπωση λοιπόν αυτή μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα αν ασκείται κριτική στην κυβέρνηση. Και αυτό είναι αρκετά ασαφές, διότι υπάρχει και εύλογη κριτική. Μετά, έχουμε την κατάσταση των ε, εργαζομένων, των μεταναστών εργαζομένων στο Κατάρ. Το 80% του πληθυσμού του Κατάρ είναι μετανάστες οι οποίοι εργάζονται εκεί και πολλές φορές αποτελούν θύματα εκμετάλλευσης. Υπάρχει απαγόρευση του συνδικαλισμού, απασχόληση με χορηγίες και αυτό καθιστά πολύ δύσκολο να παραμείνουν εκεί οι εργαζόμενοι. Επίσης, γίνεται σε τακτικά διαστήματα κατάσχεση των διαβατηρίων των εργαζομένων αυτών. Το 2022, στο Κατάρ, θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. και έχουν πολλά κατασκευαστικά έργα, έχουν αναλάβει πολλά, τους εύχομαι καλή τύχη. Υπάρχουν όμως πολλοί εργαζόμενοι μετανάστες εκεί. Αυτά λοιπόν από δική μας πλευράς, από πλευράς ανθρωπινών δικαιωμάτων, ε, ρίχνοντας μια ματιά στην κατάσταση ανθρωπινών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας, του Κατάρ και τώρα. Έχουν πάρα πολλούς συναδέλφους που λείπουν γιατί είναι στη συνεδρίαση της ΑΦΕΤ ε, βέβαια, ε, εκεί έχουν ε, άλλα ζητήματα. Για να ρίξουμε μια ματιά το τι γίνεται στο Μαγρέμπι σε άλλου χώρε, μπορούμε να δούμε ότι έχει ενεργή, ενεργή δυναμική πολιτική το Κατάρ εξωτερική. Ε, και επίσης, σε επαφές μας με τους εκπροσώπους της χώρας, να μας πούν τι, τι θα κάνουν. Ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης είναι εδώ. από το Δεν ξέρω ακριβώς ε, την ιδιότητά σας, αν θέλετε πέστε μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αν δεν έχετε αντιρρήσει να δώσω ε, το λόγο στους ε, συναδέλφους από ένα άλλο τμήμα που θα μας εξηγήσει τι γίνεται με τον ποιητή και εγώ να σας πω για τα μέσα ενημέρωση και για τους ξένους εργαζομένους, ξένους εργάτες. Ε, ευχαριστούμε που συζητάτε το Κατάρ και χαιρετίζουμε πάρα πολύ το γεγονός ότι εμείς ως ΕΕΣ και εμείς ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ε, σχολιάσουμε το τι γίνεται στη χώρα. Πρώτα-πρώτα να σας πω ότι αν και έχουμε κάποιες, ε, κάποιους περιορισμούς όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα, το Κατάρ έχει κάνει κάποια θετικά βήματα όσον αφορά το να απολάβει ο κόσμος τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η χώρα έχει θεσπίσει ένα νέο σύνταγμα εκεί όπου οι σχετικές διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, από το 2005 και μετά είναι βελτιωμένες επίσης. Είναι θετική εξέλιξη ότι η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, εκεί ε, ως παρατηρητήριο ε, ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και βέβαια έτσι είναι εδώ κανείς να κρίνει το τι γίνεται εκεί και μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα το νόμο για τα μέσα ενημέρωσης παρά τα όσα έχουν πει είναι από το 79 το 8ο σχετικό νομοθέτημα το οποίο έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση αλλά ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Έχουμε τον Υπουργό Εθνική οικονομία και πολιτισμού που πέρυσι είχε πει ότι πρόκειται σύντομα να τεθεί σε ισχύ αυτό ο νόμος και θα επικεντρώσουν την προσοχή του στην ελευθερία λόγου, θα καλύψουν όλες τις δραστηριότητε, ε, τα, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, σύμφωνα με αυτόν τον νόμο δεν θα φυλακίζουν δημοσιογράφοι, δικαστέ θα έχουν την τελευταία λέξη για όλες τις υποθέσεις που αφορούν τους δημοσιογράφους και θεωρούμε ότι και τα κοινωνικά δίκτυα θα υπαχθούν εκεί επίσης και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου όπως μπόρεσε για την προσωπία μας να, να, να ενημερωθεί δεν θα πρέπει οι δημοσιογράφοι να επικρίνουν τις φιλικές προς τη χώρα άλλες χώρες και επίσης να μην επικρίνουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας Τώρα το θέμα είναι, όπως είπατε και εσείς, τι ορίζεται μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ε, επίσης, από πληροφορίε, η Επιτροπή Σώρας έχει καλέσει όλους τους ε, ε συντάκτε, τέλος πάντων εκδότες, διευθυντές εφημερίδων για να υποβάλουν τα σχόλιά τους και αυτό το συμβουλευτικό σώμα επίσης δήλωσε ότι χρειάζεται άλλος νόμος για το διαδίκτυο και για τα κοινωνικά δίκτυα οι διευθυντές των εφημερίδων ζήτησαν από αυτό το σώμα να ε, συμφωνήσει μαζί τους όσον αφορά την ε, δίκη προσώπων που έχουν παραμεθεί σε δικαστήριο σύμφωνα με αυτό το νόμο. Τον Αύγουστο του 2012 το Υπουργικό Συμβούλιο πρότεινε να γίνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο για τα ε, μέσα ενημέρωσης κατόπιν αυτών των ε, προτάσεων του Συμβουλίου ΣΟΡΑ. ε, είναι οι τελευταίες ε, πληροφορίε που έχουμε. Όσον τώρα τους εργαζομένους, τους ελοδαπούς, για μας είναι θέμα προτεραιότητα, διότι αυτοί οι αλλοδαποί είναι το 80% του πληθυσμού του Κατάρ και επομένω είναι σαφές ότι δεν απολαμβάνουν των δικαιωμάτων οι αλλοδαποί εργαζόμενοι όπως οι υπήκοοι της χώρας. Γιατί εξαρτώνται 100% από τον εργοδότη του. Το σύστημα αυτό βελτιώθηκε κάπω, αλλά όχι αρκετά. Για παράδειγμα θα πρέπει οι εργοδότε να συνενέσουν πριν δοθεί άδεια εξόδου από τη χώρα σε οποιοδήποτε εργαζόμενο. Αλλά θα πω. Όμω, ήταν θετική εξέλιξη το γεγονό ότι τον Φεβρουάριο του 9 είχαμε ένα καινούριο νόμο που απαγορεύει το να κατακρατηθούν από τον ε, εργοδότη το αγιοσυντικά έγγραφε το διαβατήριο. Χρειάζεται δικαστική απόφαση για να μην επιτραπείς κάποιον να φύγει. Άρα χρειάζεται περισσότερη ευελιξία και αυτό το σύστημα θα αλλάξει στο εγγύ μέλλον. Η δε δραστηριότητα η σχετική τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έντονη. Έχουμε στενή επαφή με τι αρχέ τη χώρα και του βοηθούμε τόσο ώστε να βελτιώσουν αυτό το σύστημα, τόσο ό,τι ισχύει για τους αλλοδαπούς. Το ΔΕ Συμβούλιο των είχε δημοσιεύσει κάποιο φυλάδιο για, τα, για, για, τους ξένους με, με δικαιώματα και υποχρεώσεις και το Υπουργείο Εργασία διένυμε στου ξένου εργαζομένου αυτά τα φυλάδια. Έχουν δικαίωμα να απεργήσουν αυτοί οι εργαζομένοι αλλά περιορισμένο δικαίωμα απεργία. Τώρα, για του υπηκόρου τη χώρα. Δεν προστατεύονται. Πολλές φορές δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και πολλές φορές ε, φύσανται κακοποίηση σωματική και πνευματική. Υπάρχουν ε, κάποια ε, ασφαλή καταφύγια από τις πρεσβείες και έχουμε 600-700 καταγγελίες συνέχεια κάθε χρόνο για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι περισσότερε, από αυτές τι περιπτώσει καταπάτηση δικαιωμάτων αφορούν τις, τα, τα αιτήματα αλλαγής αυτού του συστήματο στη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διτή προσέγγιση όσον αφορά αυτού τους αλλοδαπούς εργαζόμενου. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να βελτιωθεί η κατάσταση των υπηκών των χωρών ε, μελών της Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τους άλλους αλλοδαπού εργαζομένου, από χώρε φτωχέ, έχουμε τακτές επαφές με τις πρεσβείες εκείνων των ε, χωρών. Προσπαθούμε δε. Να έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες και σε συνεννόηση με τις αρχές της χώρας να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την άδεια σας τώρα. Θα δώσω στον κύριο Σοπέν εδώ τον ε, διτητή Σκητάλη. Thank you, Madam uh, Ευχαριστώ πολύ. Ασχολούμαι με τα θέματα αυτά των, στα πλαίσια της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τον Νοέμβριο λοιπόν καταδικάστηκε σε ισόβια καταδίκη ο κύριος Αλατζάμι. Ε, θα ήθελα να πω ότι είναι ασύνηθες, μια, μια τέτοια περίπτωση σε, στο Κατάρ, δηλαδή ισόβια καταδίκη ε, με την κατηγορία ε, της προσπάθειας ε, ε, ε, αν, ε, And we, we have expressed uh, Uh, uh, Ανατροπή ε, της ε, κυβερνήσεως. Ε, γνωρίζετε πάντως ότι εμείς δεν έχουμε αντιπροσωπεία στο Κατάρ το ίδιο. Η αντιπροσωπεία μας έχει βάση στο Ριάντ. Όπως ορθώς αναφέρατε κι εσείς, οι ε, ε, συνήγοροι του κυρίου Αλατζάμι ε, κατήγγυλαν σειρά παρατυπιών. Θα υπάρξει βεβαίως και μια προσπάθεια να εφεσιβληθεί η απόφαση και ευελπιστούμε ότι η έκβαση της έφεσης θα είναι καλύτερη στο Κατάρ πρέπει να σημειώσουμε ότι ε, από το 2003 δεν έχουμε εκτέλεση θανατικής καταδίκης έστω και αν εξακολουθούν ε, να βγαίνουν κάποιες ε, αποφάσεις είχαμε επίσης για το, είχαμε θανατικές καταδίκες σε έξι εμπλεκόμενους σε αποτυχημένο πραξικόπημα ήδη το 1996 Βεβαίως ε, εμείς προσπαθούμε να ε, ε, συζητούμε όσο γίνεται συχνότερα και με κάθε ευκαιρία όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων στα οποία αναφέρθηκε και ο συνάδελφός μου προηγουμένως. Οπωσδήποτε προβλέπουμε μία επιτόπου συνάντηση στο Κατάρ δηλαδή το πρώτο εξάμεινο του 2013 και ελπίζουμε ότι ε, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα. Επίσης, ε, περί τα τέλη Απριλίου θα έχουμε μία συνάντηση με το Πολιτικό Συμβούλιο Εκπροσώπησης των Χωρών του Κόλπου στις Βρυξέλλες Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαπά. Σε συγγνώμη δεν σας ε, έδωσα το λόγο πραγματικά αναφέροντάς σας με το όνομά σας. Θέλει κανείς ε, να απαντήσει, να ερωτήσει κάτι. Ούτε εγώ δεν έχω ερωτήσεις λέει η Πρόεδρος. Επομένως ε, απλώς να θυμίσουμε ότι μιλάμε για διαφορετικές καταστάσεις σε διαφορετικές χώρες. Αλλά στην Αραβική Χερσόνησο σε κάθε περίπτωση και με μεγάλη ε, συχνότητα ανακύπτει το πρόβλημα των μεταναστών εργαζομένων. Στην ε, αρμόδια επιτροπή της ΑΦΕΤ έχουμε συζητήσει το ζήτημα αυτό, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ε, το θέμα των μεταναστών εργαζομένων μπορεί να εξεταστεί στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων και θα πρέπει ίσως να ανακύπτει το ζήτημα ε, όταν ε, παίρνουμε τις ε, γενικές κατευθύνσεις προσέγγισης της ευρύτερης περιοχής και όχι μονάχα στις διμερείς επαφές που έχουμε αναχώρα. Ε, για χώρες όπως η δική μου ο τρόπος ε, κάλυψης ε, των εργαζομένων στην Αραβική Χερσόνησο θυμίζει λίγο συνθήκες σκλαβιάς και επομένως θα πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά το ζήτημα αυτό. Πολύ ωραία. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τόιερμαν πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κόχομ, σχετικά με τις επερχόμενες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μπορείτε να έρθετε κύριε Τόιερμαν εδώ. Yeah. So, um, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τόιμαν που ξαναήρθατε στην ε, Επιτροπή μας ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε συχνή ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε ή να εντείνουμε τις εργασίες μας, ε, πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερο επίπεδο συνεννόησης και αποτελεσματικότητας στα ανθρώπινα ε, δικαιώματα και επομένως ε, για μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό να ε, ερχόμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Ε, συχνά προσκαλούμε τους αναθέμα αρμοδίους ε, για να, εδώ στις Βρυξέλλες για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί περαιτέρω να αναπτυχθεί η ατζέντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις ανακοινώσεις μου χτες είπα ότι καλωσορίζω το γεγονός ότι είπα ότι εκπρόσωπος Νάβε Πιλάη, θεωρεί ότι είναι σημαντικό και θετικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να ε, είναι ε, παρόν σε αυτήν την τεράστια εκδήλωση της Γενέβης. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ε, έχουν πολύ θετικό αντίκτυπο γιατί ε, μέσω της δράσης αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει ε, την εξέλιξη της ατζέντα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίως δεν παίρνονται οι αποφάσεις εδώ στην Επιτροπή μας αλλά και ε, ξέρουμε ότι ε, θα μπορούσαμε να είμαστε και πιο αυστηροί απέναντι και στους εαυτούς μας γιατί ξέρουμε ότι και εμείς στις δικές μας χώρες έχουμε περιθώρια βελτίωσης ε, των καταστάσεων όσον αφορά ας πούμε την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ανάδυσης των νεοναζιστικών κομμάτων και δράσεων. και επομένως καλό θα ήταν ε, να ε, μπορέσουμε να ξεπεράσουμε κάποια δικά μας προβλήματα και με τον τρόπο αυτό να γίνουμε και πιο αποτελεσματικοί σε διεθνές επίπεδο η ατζέντα των, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι πάντα πολύ συγκεκριμένη και θα θέλαμε να μας πείτε μερικά πράγματα παραπάνω για να καταλάβουμε τι θα γίνει σε αυτήν την 22η συνεδρίαση, τι θα εγγραφεί ε, στην ε, ε, ε ημερήσια διάταξη, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες για αυτή την νεαρινή συνεδρία. Ήρθατε χθες από τη Γενέβη και τα συζητήσατε όλα αυτά εμείς προτιθέμεθα να στείλουμε και αντιπροσωπεία στην Γενέβη από τις 22 Φεβρουαρίου μέχρι τις, ε, μέχρι τις αρχές Μαρτίου και θα προετοιμάσουμε μάλιστα με την ευκαιρία και ένα σχετικό ψήφισμα το οποίο 80% βέβαια στρέφεται προς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά θέλουμε να σας ακούσουμε, ενδεχομένως ε, μετά από αυτά που θα μας πείτε, να τροποποιήσουμε κάπως και το ψήφισμά μας, να προσθέσουμε κάποια πράγματα. και βεβαίως τα διάφορα θέματα και οι επιμέρους ε, καταστάσεις ανακράτος εξακολουθούν και μας ε, απασχολούν. Αλλά νομίζω ότι χθες αποφασίσατε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του Συμβουλίου. Μπορείτε να μας τις πείτε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την πρόσκληση Ήρθα για να σα ε, αναφέρω τι προτεραιότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ενδιαφέρει μόνο αυτή την Επιτροπή, αλλά γενικότερα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Ηνωμένα Έθνη. Θα γίνουν πολλές σημαντικές ε, συναντήσεις στο άμεσο μέλλον και εσείς μας είπατε ότι θα πάτε στην Γενέβη με τη δική σας αντιπροσωπεία φέτος. Και εμείς προετοιμάζουμε το χρονοδιάγραμμά μας και επίσης με χαρά μας να δούμε τα ψηφίσματά σας. Επίσης, θεωρούμε πολύ θετικό το γεγονός ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα μέσα που διαθέτουμε και είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ανακαλύψεις και τα βρήματα των εισηγητών ε, σχετικά με τις ε, εκάστοτε ε, χώρες. Χρειαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς που διαθέτουμε και να τους θέσουμε σε ισχύ. Δεν αρκεί μόνο η δέσμευση στα λόγια, χρειαζόμαστε και πράξεις. Και στο Συμβούλιο και στην Ομάδα εργασία στα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουμε καλέσει εμπειρογνώμονε και προσπαθούμε να καταρτήσουμε εκθέσεις και να αναπτύξουμε στρατηγικές ε, σχετικέ με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική κατάσταση. Για εμάς επίσης είναι σημαντική αυτή η προεργασία όταν ε, ασχολούμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορες ε, τρίτε χώρες. Τώρα, να σα μιλήσω για το 2012. Έγινε πολλή δουλειά πάνω στο στρατηγικό πλαίσιο για την ε, δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρή δέσμευση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πλήρη χρήση των ε, μέσων που διαθέτει και του συστήματος που υπάρχει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά είναι να βελτιώσουμε και να συνεισφέρουμε και να διασφαλίσουμε ότι αυτά που λαμβάνουν χώρα στην Γενέβη και στη Νέα Υόρκη υιοθετούνται και ενσωματώνονται και στην δική μας δουλειά. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε κάποιον αντιπρόσωπο στην ε, ειδική ανώτατη ομάδα στα Ηνωμένα Έθνη για να κάνουμε τις ε, θέσεις μας γνωστές, ιδιαίτερα και όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Έχουν προσκληθεί επίσης και αντιπρόσωποι πολιτικοί υπουργοί από τις χώρες με τις οποίες ασχολούμαστε για να συζητήσουμε το θέμα αλλά και για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Η δέσμευσή μας επίσης περιλαμβάνει μια πιο στρατηγική και συστηματική προετοιμασία για το 2013 για τις εργασίες μας στα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε συνεδριάσεις το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο, επιτροπές και από το 2012 αποκομίσαμε θετικές εμπειρίες από τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκαμε, από τις συμμαχίες, από τη καλή συνεργασία που καταφέραμε να έχουμε με τις τρίτες χώρες. Έγιναν σημαντικές βελτιώσεις με τις σχέσεις μας με τη Λευκορωσία, για παράδειγμα, με τον αγώνα για το μορατόριο για την ε, θανατική ποινή. Και αυτό σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε. Το σχέδιο δράσης, επομένως, τονίζει την, ε, τον καλό στρατηγικό σχεδιασμό. Πέρυσι είχαμε καλά αποτελέσματα Σχεδιάσαμε ακριβώς αυτά που θέλαμε να κάνουμε στο πρόγραμμα του 2013 και έτσι θα συνεχίσουμε και φέτος. Είναι πολύ σημαντικό στην Γενέβη να υπάρχει ένας καλός στρατηγικός σχεδιασμός και να είναι προσκεκλημένοι οι κατάλληλοι αρμόδιοι εμπειρογνώμονες. Μπορώ να σας ε, πω σήμερα ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες για τις ε, συνεδριάσεις του Μαρτίου. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι τα αποτελέσματα φυσικά, όμως σημαντικό είναι ο διάλογος με τι τρίτε χώρε. Στις 18 Φεβρουαρίου θα γίνει η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όπου θα ψηφιστούν συμπεράσματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία θα αρχίσουν να ισχύουν από το Μάρτιο και στο εξή. Επίση, να σα ενημερώσω για... θα σας ενημερώσω για τις σχετικές εκθέσεις που θα συνταχθούν. Προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο είναι να, αντιμετωπίσει την κατάσταση στην Συρία. Η Συρία είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς. Χθε στη συνάντηση που είχαμε πρώτο θέμα ήταν ανταλλαγή ε, απόψεων και πληροφοριών με την αποστολή για την Συρία. Είχαμε μια έκθεση την οποία αναφέρθηκαν τα κύρια ευρήματα, όμως πραγματικά μας ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται όσον αφορά τις ε, παραβιάσεις, τις διάφορες παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και να τονίζουμε το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει εκεί και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Ε, βέβαια, έχουμε, πολύ, έχουμε περιορισμένα μέσα, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο Ανθρωπίων Δικαιωμάτων, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε την εργασία μας, πρέπει να επεκταθούν οι αρμοδιότητές μας και ταυτόχρονα να συνεχίσουν οι εκθέσεις και η τακτική πληροφόρηση, έτσι ώστε να είμαστε πάντα ενήμεροι για τις ε, νεότερες εξελίξεις και ίσως μπορέσουμε για πρώτη φορά να υιοθετήσουμε με ομοφωνία συμπεράσματα για την κατάσταση στη Συρία. Η τωρινή σύνθεση του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή εργάζεται προς την δημοσίευση μιας ανακοίνωσης ενός μηνύματος που θα αναφέρεται στην ε, λογοδοσία και ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντομα. Θα συνεργαστούμε πολύ στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τουρκία και ορισμένες ε, αραβικές χώρες ε, του Αραβικού Συνδέσμου προς το στόχο αυτό. Επίση, σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη και θέμα για το οποίο έχουν ήδη αρχίσει διαβουλεύσει είναι η κατάσταση στη Μιανμάρ. Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει δραματικές εξελίξεις και έχουμε πολλές ανησυχίες για τους πολιτικούς κρατούμενους. Και, για, και εκτός από αυτό για πάρα πολλά θέματα ακόμα. Υπάρχει ε, μια αντιπροσωπεία που σκοπεύουμε να στείλουμε και να συνεργαστούμε με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι μια δέσμευση για υπογραφή μνημονίου συνεννόησης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον ε, ύπατο αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. μνημόνιο και για συνεχής επιτήρηση της κατάστασης αλλά και για αποστολή ε, τεχνικής βοήθειας διότι χρειάζεται να βελτιώσουμε και να εμπλουτίσουμε το υπάρχον μνημόνιο συνεννόησης του Συμβουλίου. Επίσης, άλλα σημαντικά θέματα. Η Βόρεια Κορέα πρέπει να ανανεωθεί η εντολή του ειδικού εισηγητή, αλλά και υπάρχει ανάγκη να βρεθούν νέες στρατηγικές ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων. Με τα στρατόπεδα φυλακισμένων, με τις απαγωγές, Αυτή τη στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένε Πολιτείες, την ε, Ιαπωνία για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και σκοπεύουμε να διεξάγουμε εκθέσεις ε, εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει την ε, πρόταση να ανανεωθεί η εντολή του αρμόδιου για τα ζητήματα στην περιοχή αυτή. Το γραφείο του ΙΠΑ του Αρμοστή έχει επίσης δημοσιεύσει πρόσφατα ανακοίνωση για τα γεγονότα στο Μάλι. Υπάρχουν βέβαια και άλλα ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά να σας πω ότι τον Ιούνιο το ε, κύριο θέμα για μας θα είναι η κατάσταση στη Λευκορωσία, το Σεπτέμβριο Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Ερυθρέα, Καμπότζη, Βόρεια Κορέα. Ελπίζουμε και το Μάρτιο να καταφέρουμε να φέρουμε στην ημερήσια διάταξη την Βόρεια Κορέα. καθώς και η ανανέωση της εντολής του ειδικού εισηγητή για την ελευθερία θρησκείας και πεπιθήσεων. Θα παρουσιάσουμε ένα ψήφισμα επίσης για τα δικαιώματα του παιδιού και θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα, τα δικαιώματα των γυναικών για παράδειγμα, την ισότητα των ε, φύλων, την βία ε, ενάντια στις γυναίκες. Δεν θα είναι προτεραιότητα μόνο το Μάρτιο, αλλά και θα συνεχιστούν και μετά από αυτόν. Όσον αφορά για τη βία ενάντια στις γυναίκες, αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε και προσπαθούμε να συντάξουμε μία ανακοίνωση και να εμπλουτίσουμε την, ε, το ψήφισμα του Συμβουλίου. Τώρα, όσον αφορά τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των Ηνωμένων Εθνών και την πρόσβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, προσπαθούμε να πιέσουμε, διότι πολλές φορές οι χώρες χρησιμοποιούν αντίπεινα, χρησιμοποιούν εκβιασμό, εκφοβισμό προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτές τις χώρες η... το πεδίο δράσης των μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ολαιόνα και συγκνώνεται. Μια άλλη διαδικασία θα είναι η διαδικασία δηλαδή θα γίνει μεταρρύθμιση του στήματος του ΟΗΕ. Πρώτη για μια διαδικασία διαπραγματεύσεων θα γίνει στη Νέα Υόρκη, αλλά είναι πολύ σημαντική γιατί για τα ανεξάρτητα παρατηρητήρια είναι η καρδιά του συστήματος. Θα πρέπει να περισσοθεί, είναι τεράστιες οι προκλήσεις και πολιτικά και οικονομικά. Ο... Βέβαια, θα πρέπει να κυρώσουν τη συνθήκη πολλά κράτη για να το σύστημα και πρέπει θέλουμε του υπάτου εκπροσώπου την ανεξαρτησία και θέλουμε επίσης η παγκοσμιότητα των ανθρωπινών δικαιωμάτων επίσης να περισσοθεί γιατί εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε καλά για αυτές τις συζητήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Τόρμαν. Είναι πολύ σαφές τώρα το τι θα είναι σήμερα στη διάταξη και τώρα ήρθε η ώρα οι συνάδελφοι να άλλων παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Κυρία Ντεκάιζερ, νομίζω πάρα πολύ συχνά έχετε ασχοληθεί σε επίπεδο ΟΗΕ με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ. Κύριε, για όλα όσα μας εξηγήσατε. Είναι αλήθεια και γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ΟΗΕ το έργο που επιτελείται είναι θαυμάσιο. Μας περιγράψετε το τοπίο με πληρότητα. Εμείς θα επιτόπου με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε έχουμε τα θεσμικά ζητήματα από την μια μεριά και από την άλλη έχουμε την ομή πραγματικότητα που πολλές φορές απέχει πολύ το ένα από το άλλο. Θα σταθώ σε δύο-τρία σημεία για να δούμε τι μπορείτε να κάνετε. Πρώτα πρώτα, πρόσφατα, είχαμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από πλευράς Ελβετίας, αφορά τη Συρία, γιατί έχει ζητηθεί να ασχοληθούμε με τη χώρα εκείνη και τη Συρία. Αν θυμάμαι καλά, η Ελβετία το Λουξεμβούργο, αν θυμάμαι καλά, η Μεγάλη Βρετανία, η Κορέα, κάποιες χώρες ενέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία για τη Συρία. Και δεν μπορώ να διαπιστώσω ακριβώς αν έχει τον πρωτονιστικό ρόλο που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό με πειράζει. Μας μιλήσατε για τη Συρία, για ότι χρειάζεται να γίνει έρευνα εκεί. Γιατί όμως εμείς που έχουμε τόσα θεσμικά όργανα δεν έχουν προβληθεί στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας παρά τις ε, γνωστές δυσκολίες σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας ξέρουμε ποια είναι η ισορροπία δυναμική ε, όμως πρόκειται για μια προβεβλημένη πολύ σημαντική πρωτοβουλία ακόμα ε, είμαστε στα παρασκήνια Κάτι άλλο τώρα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει, οπωσδήποτε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα, θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι στην καρδιά της πολιτικής που ασκούμε και όσον αφορά τη Συρία. Βλέπουμε τι διαδραματίζεται εκεί. Βέβαια υπάρχουν και τα θέματα τα δημισιονομικά σε επίπεδο συμβουλίου αλλά η ανθρωπιστική βοήθεια είναι κάτι το οποίο είναι δυνατόν να παρασχεθεί στους ίδιους πρόσφυγες. Είναι θέμα ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αφορά το Συμβούλιο, αφορά τον προπολογισμό. Εν κενό λειτουργείτε ή τέλο πάντων έχετε κάποιο είδους ε, δυνατότητα να επηρεάσετε το Συμβούλιο για τα θέματα αυτά που τελικά είναι θέματα σύνδεξη Λισαβόνα. Είναι αυτά τα δύο ζητήματα που νομίζω ότι με απασχολούν, με πάρα πολύ και αφορούν τη Συρία. Κάτι άλλο τώρα, και εκεί θα βάλω τελεία για να μιλήσει άλλο συνάδελφο, είναι κάτι το οποίο αφορά άμεσα αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη. Και ενώ τις χώρες όπου έχουμε κάποιες εκτροπές σε επίπεδο των δικαιωμάτων. Λέμε δεν είμαστε στο Κονγκό, είμαστε στη Συρία. Αλλά α, πριν από λίγο ήμουν στην ε, Αίγυπτο και προβληματίζομαι για αυτή τη διαγραφή του, του άρθρου που αφορούσε δικαιώματα, τα, τα δικαιώματα των γυναικών. Ε, καταργήθηκε το άρθρο το οποίο ε, αφορά κάποια εγκλήματα που γίνεται κατά τη ευθεία έκφραση, κάτι που θεωρούνται. Ε, κάτι που δεν μπορεί να πει πράγματα θεωρούνται βλασφημία και τους βιασμούς των γυναικών και τελικά πρόκειται πολύ σοβαρά γεγονότα αλλά δεν είδα να αντιδράσαμε συζητούμε εδώ στο κοινοβούλιο αλλά ίσως θα πρέπει να προσέξουμε για αυτά τα λογιστήματα τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους σοβαρούς να τρώμε δικαιώματα αυτά. Πάντως, ξέρετε ότι στηρίζουμε το έργο σας και η συνεργασία μας είναι πάντοτε εργαστή. Ευχαριστώ κύριε Ντεκάζη. Δεν βλέπω άλλους να ζητούν το λόγο. Έχω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις, ίσως τις απαντήσετε από κοινού. Αναφερθήκατε στις διάφορες προτεραιότητες. Πρέπει να σας πω ότι όλες αυτές οι προτεραιότητες σχετίζονται και με την εργασία που κάνουμε εμείς. Ας πούμε, εμείς αποφασίζουμε ε, να ε, και η δική μας Επιτροπή και η ΑΦΕΤ ε, να ε, πάρει, να κάνει ψηφίσματα ε, όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες ε, και την πτυχή που περιλαμβάνουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. And uh, we will send delegation most likely in May. όσον αφορά την Μπούρμα και τη Μιανμάρ, για τον Μάρτιο, το Μάιο είπαμε ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό η συμφωνία ε, ε, να ανοίξει ε, στην Κανκούν ένα γραφείο νομίζω ότι είναι σοφή απόφαση και σχετίζεται βεβαίως και με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δίνουμε 4 εκατομμύρια στο γραφείο του, του, της ΥΠΑ του Αρμοστού και ε, ε, διαρκώς εκείνη αναφέρει παραπάνω εργασίες και βεβαίως ε, το άνοιγμα ενός field office θέλει στήριξη και θέλει και χρηματοδότηση. Όσον αφορά τη Βόρεια Κορέα, είχαμε την προηγούμενη χρονιά ακρόαση. Η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ καλή και ελπίζουμε ότι εάν υπήρχε μια ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας ε, θα βοηθούσε και το ίδιο το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και για τις γειτονικές χώρες. Πρέπει είναι καλό που μπαίνει στη μέση διάταξη. Τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει ε, να ασχοληθούν και με το θέμα αυτό. και ελπίζω να αποφασιστεί κάποια στιγμή γιατί θα ήταν εξαιρετικό να έχουμε μια επιτροπή διερευνητική επί των θεματικών τώρα ε, στοιχείων. Σήμερα το πρωί αποφασίσαμε ότι η Επιτροπή μας θα κάνει έκθεση σχετικά με τις νέες κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, για την ελευθερία θρησκευτικών και λοιπόν πεπιθήσεων. Επίσης θα επιμηκυνθεί η εργασία του ειδικού εκπροσώπου για τα ίδια θέματα. Ε, αρκετές ε, χώρες έχουν ε, θεωρήσει ότι δεν είναι καλή η θητεία του ή η εντολή του δεν είναι αντικειμενική. Είναι σωστό λοιπόν να τον στηρίξουμε. Βεβαίως και το θέμα των ΛΟΑΔ είναι πολύ σημαντικό είναι κάτι που επανέρχεται από πολλούς βουλευτές και σε πολλές επιτροπές οι οποίες ε, ε, ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια άλλη χώρα ή θέμα, όμως το ψήφισμά μας ε, θα δείτε ότι είναι αρκετά ε, έτσι, διευρυμένο ε, και είπαμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε και πιο πολύ όσον αφορά την Σρι Λάνκα και να στηρίξουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι σημαντικό ζήτημα. Όμως δεν άκουσα τις πολιτικές ομάδες ε, εάν υπάρχει κάποια χώρα άλλη πέρα από αυτές που αναφέρατε που θα πρέπει να προσθεθεί στο ψήφισμά μας, αλλά αυτό θα το δούμε και αργότερα. Και επίσης, να πω σε όλους σας, ε, όταν ε, ταξιδεύουμε σαν αντιπροσωπείες, ε, βλέπουμε ότι η εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ δραστήρια και οργανώνει ε, συναντήσεις ε, με τους πρέσβεις των χωρών κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ορισμένες χώρες εμποδίζουν κατά κάποιο τρόπο την εργασία της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη ΣΥΠΑ ή ε, στην Γενέβη γιατί αρχίζουν και λένε «Μα αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα, α, πρέπει να διαβουλευτούμε μεταξύ μας». Ε, και αυτό δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνους και προσπαθούν μάλιστα να επηρεάσουν και άλλα μέλη λοιπόν και έχουμε και κάτι άλλο ένα άλλο βράδυ που θα είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να καλέσουμε ε, τους ε, πρέσβεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φορά που γίνεται αυτό, εγώ βέβαια ήμουν παρούσα μία φορά μόνο, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι κάθε φορά είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εκεί μπορεί κανείς να συζητήσει για μερικές καθολικές ανθρωπιστικές αξίες και μπορούμε να συζητήσουμε για τον Μπαχρέιν, για την Αιθιοπία. Ε, είναι καλό να καλέσουμε δηλαδή και τους εκπροσώπους σε τέτοιων χωρών έτσι ώστε να δούμε πώς βλέπουν εκείνη τη δουλειά του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στη συνάδελφο, να κάνει την ερώτησή της και μετά να απαντήσετε σε όλους μαζί. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Λεζέρ. Δυστυχώς οι διερμηνείς δεν ακούν. Δυστυχώς οι διερμηνείς εξακολουθούν να μην ακούν. Ωραία, τώρα άνοιξε το μικρόφωνο μου, λέει η κυρία Λουζέρε. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές ασυνάπειες, ασυνέπειες της Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά και την εξωτερική πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι συζητήσεις που γίνονται στα Ηνωμένα Έθνη νομίζω ότι απεικονίζουν πλήρως την κατάσταση. Κοιτάξτε, εγώ έχω μια αιμονή, όπως αρκετή μεταξύ ημών. Η εμπονή μου λοιπόν είναι η Τουρκία και η ειρηνευτική διαδικασία στην ε, Τουρκία. Ε, εγώ είμαι Γαλλίδα και είχαμε πρόσφατα τρομερές δολοφονίες ε, στην, στην γαλλική επικράτεια. Επομένως θα πρέπει πέρα από οποιασδήποτε προσπάθειες παγίδευσης ή χειραγώγησης θα πρέπει να δούμε την κατάσταση και θα πρέπει όλοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη να βάλουν το λιθαράκι τους έτσι ώστε να βοηθήσουμε πράγματι την Τουρκία. 30 χρόνια πόλεμο, 45.000 έχουν ε, απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Νομίζω ότι είναι αρκετά. Δεν χρειάζεται να έχουμε και άλλα θύματα. Βλέποντας να δούμε από κοντά την Τουρκία και κυρίως την κατάσταση των μειονοτήτων στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ναι, ίσως και εσείς κύριε Τόιρμαν θα μπορούσατε να πείτε δύο λόγια πάνω σε αυτό. Την προηγούμενη φορά είχαμε ε, μία σειρά συναντήσεων μεταξύ αυτών και με τον ε, πρέσβη του ε, Ισραήλ που παραπονέθηκε ισχυρότατα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη χώρα του η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη και αυτά. Ακούω φήμες ότι ενδεχομένως το Ισραήλ ε, προσανατολίζεται ε, να μην ακολουθήσει τις συστάσεις της Universal Periodic Review. Αυτό θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνεται και νομίζω ότι θα δυναμητήσει την ίδια τη λειτουργία του συστήματος. Για πέστε μας κάτι γι' αυτό. Um, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για τις ερωτήσεις σας. Δεν είμαι αρμόδιος για να απαντήσω σε όλες, αλλά θα προσπαθήσω όσο καλύτερα μπορώ. Όσο για τη σχετικότητα των συζητήσεων στη Γενέβη και για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχέσεις μας γενικότερα. Παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια την δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ και έχω μία εικόνα του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα πιστεύω πως έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος. Όντως, στο παρελθόν είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι η Γενέβη ζούσε σε μία φούσκα και ό,τι γινόταν εκεί, τα θέματα τα οποία συζητούσαν δεν ε, ενσωματώνονταν στην ε, δική μας ε, πολιτική. Υπήρχε εντύπωση ότι δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε τους στόχους μας στην Γενέβη διότι δεν είχαμε υποστήριξη, διότι δεν το είχαμε συζητήσει ανοιχτά αλλά διμερώς και θα ήμασταν πιο αποτελεσματικοί εάν εκτός από τις συζητήσεις στη Γενέβη έχουμε και πολιτικούς διαλόγους και διμερείς ε, συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, αλλά εκτός από αυτό και να συνδέσουμε καλύτερα αυτά που γίνονται εκεί με, την, ε, με εμάς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει καλύτερο στρατηγικός σχεδιασμός και συνεργασία. Αυτό που κάνουμε στη Γενέβη είναι ένα μέρος της γενικής ε, συνολικής μας στρατηγικής. Και αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση της ε, ε, Μιανμάρ. Συνεργαζόμαστε στενά για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής. Αυτό κάνουμε και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίπτωση της ε, Συρίας. Συνδέεται η δουλειά μας για τη Συρία με τη γενική μας πολιτική για το θέμα. Αναφερθήκατε στην ελβετική επιστολή του ε, Ελβετού πρέσβη στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εκ μέρους 55-56 διαφορετικών ε, κρατών που, το, που υπέγραψαν την επιστολή αυτή. Να σας πω ότι 26 κρατή την υπέγραψαν την επιστολή αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν ε, αναφέρουμε την κατάσταση στη Συρία, είτε είναι κάποιος υπουργό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται πάντα το ζήτημα της λογοδοσίας. Το Δεκέμβρη ιδιαίτερα τονίστηκε από το Συμβούλιο η υποχρέωση λογοδοσίας και έγινε έκκληση στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στο Διεθνές Δικαστήριο να ασχοληθούν εντονότερα με το θέμα και να ακολουθήσουν τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί. Φυσικά, το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί και στη Γενέβη. Και βέβαια, προσπαθούμε και τη συνεχίζουμε να προσπαθούμε να αυξήσουμε την, την, ε, τις πολιτικές δεσμεύσεις ενασχόλησης με την Συρία και να συνδέσουμε καλύτερα τις εργασίες μας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας και ο κύριος Πινιέρο ε, τόνισε την ε, θετική του άποψη για την ε, συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την ε, Μιανμάρ τώρα, έχουμε πολλές προκλήσεις. Η κύρια πρόκληση είναι η συνεργασία και ο προϋπολογισμός ο οποίος έχει μείνει δεν έχουν αυξηθεί τα κονδύλια Και συνάδελφοι στην χθεσινή συνάντηση από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ συναντήθηκαν, συζητήσαμε μαζί τους και τους είπαμε ότι εκτός από τα υπάρχοντα κονδύλια που απευθύνονται στην ε, Μιανμάρ έχουν αποδεσμευτεί και 4-5 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ. Προσπαθούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν επαρκέστερη στήριξη για την δουλειά που κάνουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Ηνωμένα Έθνη. Όσον αφορά τη Βόρεια Κορέα, υπάρχει μια γενική συμφωνία για την ανάγκη να προχωρήσουμε παραπέρα. Βέβαια η δουλειά του αρμόδιου εισηγητή είναι εξαιρετική, όμως χρειαζόμαστε περισσότερα, χρειαζόμαστε ένα ανεξάρτητο όργανο που θα συνεισφέρει περισσότερο στην ε, θετική έκβαση της υπόθεσης. Επίσης, όσον αφορά την, ε, του Συμβουλίου Ελευθερίας Θρησκείας και Πεπιθήσεων, και εκεί υπάρχει βελτίωση Υπήρχε μια έκθεση στην ε, Γενική Συνέλευση όσον αφορά την, ε, τον προσιλητισμό όπου αναφέρθηκε έντονα το δικαίωμα του να αλλάξει κάποιος τη θρησκεία και τις πεπιθήσεις του και αυτό είναι μέρος της ελευθερίας ε, θρησκείας και πεπιθήσεων. Επίσης, ο δικό ε, εισηγητή να πω ότι μέσω των εκθέσεών του συνεισφέρει στην πρόθεση του ζητήματος. Τέλος, Τουρκία. κυρία Βερσόν αναφέρθηκε σε αυτό. Να απαντήσω και να πω ότι βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θίγει κάθε θέμα ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών. Προσπαθεί να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και με την Τουρκία υπάρχουν και άλλες ε, οδοί επίλυσης ε, από το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχει, υπάρχουν περιοδικές εκθέσεις, έχουμε όργανα με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, υπάρχουν ευρήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε διμερώς με την Τουρκία. Και τέλος, κυρία Μπίλερ, Ισραήλ, να σας πω το εξής. Ε, το Ισραήλ δεν ήταν πλήρε μέλο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όμω έχετε δίκιο. Τον τελευταίο Απρίλιο έστειλε το Ισραήλ μια επιστολή στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στον ΙΠΑ το αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην οποία δήλωσε πως αποχωρούν και κατέστη σαφές ότι το Ισραήλ πλέον δεν θα συμμετέχει στην περιοδική έκθεση. Δυστυχώς αυτό. Είμαστε της άποψης ότι όλα τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να συνεργαστούν για τη βελτίωση των μηχανισμών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι το Ισραήλ αισθάνεται απομονωμένο λόγω της ε, κατάστασης και αυτό χρήζει συζητήσεων από την άλλη, η περιοδική έκθεση έχει ως κύριο θέμα την ίση αντιμετώπιση όλων των χωρών, είτε του Ισραήλ, είτε των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Γαλλίας. Όλες οι χώρες δηλαδή να γίνονται αντικείμενο τακτικής εξέτασης από την περιοδική έκθεση. Εμείς αποφασίσαμε να ε, Εμείς ε, θεωρούμε το ότι η απόφαση του Ισραήλ να μην συμμετέχει είναι πολύ αρνητική και για το ίδιο το Συμβούλιο, αλλά και πιστεύουμε ότι δεν είναι καλό και για το ίδιο το Ισραήλ. Δεν θα το ωφελήσει. Αυτές τις, ε, αυτές τις μέρες στη Γενέβη προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση για αυτό το θέμα. Και το μόνο θετικό ήταν τουλάχιστον ότι το Ισραήλ ζήτησε μία αναβολή τη συζήτηση ε, του θέματο. Όμω, μέσα στο 2013 το Ισραήλ θα εξεταστεί από την περιοδική έκθεση. Σα ευχαριστούμε για το όνομα, Πρόεδρο. Τέλειωσε ο χρόνο που είχαμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα και σίγουρα πρόκειται να έρθουμε σε επαφή μαζί για να προετοιμάσουμε τι λεπτομέρειε τη επίσκεψη. Τώρα, φτάνουμε στο τελευταίο θέμα τη ημερησία διατάξεω. Ο κ έχει ζητήσει να εξετάσουμε την κατάσταση στο Καζακστάν και πάλι κάτι το οποίο μας είχε απασχολήσει τακτικά και έχουμε και την κυρία Νίλσεν που είναι η εισηγήτρια της ε, ΑΦΕΤ και θα δούμε τις επιδόσεις της χώρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έχουμε από την υπηρεσία εξωτερική δράση. Ποιον έχουμε, ποιο είναι. Ε, πάντοτε τη την στη διάταξη. Θα θέλαμε τουλάχιστον μία μέρα πριν να ξέρουμε ποιο πρόκειται να μα επισκεφθεί. Ούτω ώστε με την δέουσα ευγένεια να μπορώ να σα παρουσιάσω και να αναγγείλω το όνομά σα. Be um, good uh, if you you start with your impact to update us on the. Οπότε παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την κατάσταση στο Καζακστάν. Διότι το Νοέμβριο... Α, καλά, τέλος πάντων. Καλά, να μην, να μην πω αυτό που θα πείτε κι εσείς. Um, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ασχολούμαι στην εξωτερική υπηρεσία εξωτερικής δράσης με το Καζακστάν. Συγγνώμη που δεν σας ε, παρουσιάσαμε πριν ποιος θα έρθει και στην Επιτροπή μας έχουμε συζητήσει και είπαμε ότι έχουμε προβληματιστεί, ανησυχούμε από τότε που δικάστηκαν εκείνοι οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια τον Ιούνιο. Επίσης πέρασε από δικαστήριο ο κύριος Κοσλόφ τον Οκτώβριο που είναι ο, ένας από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Υπήρξε μια πρωτοβουλία του ε, αρχής Αγγελέως. Είχαμε... Ε, τέλος πάντων προσπάθησαν να φημώσουν πολλές εφημερίδες και διάφορα websites. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι καλύπτανε τρομοκρατικέ ενέργειες και έτσι ε, απειγόρευσαν την κυκλοφορία των εφημερίδων και έκλεισαν αυτά τα site. Το Νοέμβριο λοιπόν έγινε και μια επίσκεψη, είχαμε τότε και υπουργική συνάντηση για την ε, ασιατική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μπισκέκ, επομένως πήγαμε εκεί και είδαμε τον Ναζαρμπάγεφ και οι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος πάντων συζήτησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα επίσης στο Πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας του Καζακστάν, του Αζερμπαϊτζάν. Ε, έγινε μια διάλεξη για αυτά τα ζητήματα γιατί από την αρχή είχαμε αυτή την πολιτική και είχαν γίνει από την κυρία Άστον δηλώσεις όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εμπορικές ε, σχέσεις και είπαμε να γίνει μια καινούργια συμφωνία συνεργασίας η οποία θα θέλουμε να εξαρτάται από το τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πολιτική δεν έχει αλλάξει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν αυτών, όπως εσείς έχετε ξαναπεί εδώ, μετά από τη συνάντηση του Καζακστάν της ε, Διακοινοβουλευτική Επιτροπής και κατόπιν που είχαμε στην ΑΦΕΤ την, ε, την Τρίτη ε, τη συνάντηση με την αντίστοιχη ε, αντιπροσωπεία και είχαμε επίσης στις 22 Νοεμβρίου ένα ψήφισμα και είπαμε ότι είναι πολύ σημαντική η χώρα του Καζακστάν από πλευρά εμπορίου, πλευρά ενεργεία και επίση είναι σημαντικό παράγοντα στην περιοχή. Και κατόπιν είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε σχέσει σφαιρικέ για όλα, αλλά πρέπει οι προβληματισμοί, τα ενισχύσει με τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να, να, είναι προπόθεση για τι υπόλοιπε σχέσει. Και είπατε εκπρόσωπο και σχετικές υπηρεσίες είπαν ότι η εξελίξη των τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σχετικές εξελίξεις και σε σχέση με, με την αντιπολίτευση και σε σχέση με τον κύριο νόμο για την θρησκεία, για τις ε, θρησκευτικές μειονότητες στο Καζακστάν και όλα αυτά τα αναδεικνύουμε στην ανακοίνωσή μας και τα αναφέρουμε με τους, τους συνομιλητές μας από το Καζακστάν κάθε φορά και παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά. Ευχαριστούμε κύριε Βεζιά. Νομίζω ότι το γεγονός ότι εξακολουθείτε να ασχολείστε με το θέμα του Καζακστάν που παίζει ρόλο σταθεροποιητικό στην περιοχή είναι πολύ σημαντικό. Εάν ε, βλέπουμε μια κατάσταση όπου ας πούμε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης ε, φυλακίζεται για 7 χρόνια ή τέλος πάντων εκδίδεται εναντίον του δικαστική απόφαση για επταετή εγκλισμό ε, αυτό προφανώς ε, θα αποβεί αποσταθεροποιητικά το Καζακστάν ε, είναι και μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και επομένως ε, αργότερα στην Γενέβη ε, ενδεχομένως θα μπορέσουμε να συναντήσουμε τον πρέσβη του Καζακστάν έτσι ώστε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Και άλλωστε για να εκλεγεί κανείς αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει καλό μητρό και καλά αποτέλεσμα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, Νέλσαν, Νέλσον, ευχαριστώ πολύ. Επανειλημμένα βεβαίω έχω εκφραστεί επί του θέματο, δηλαδή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν. Ε, εδώ και ένα χρόνο ο Βαζιμίρ ε, Κοσλόφ βρίσκεται στη φυλακή οι Ευρωπαίοι και όλοι οι εκπρόσωποι της κοινότητας που ήταν παρόντες στην δίκη είπαν ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία έτσι ώστε να καταδικαστεί σε 7 χρονη φυλάκιση πέρα από την απόφαση της κασακικής κυβερνήσεως να φημώσει μέσα ενημέρωση, να καταφερθεί εναντίον της ελευθεροτυπίας κτλ αυτά που συμβαίνουν στο Καζακστάν κατά την άποψή μου είναι σοβαρά ε, και όπως λέει και η κυρία Άστον πολύ συχνά με απασχολεί, προβληματίζομαι, καλό είναι αυτό αλλά δεν αρκεί ε, το να εκφράσει κανείς τον προβληματισμό του αλλά ε, να αφήνει την κατάσταση να επιδεινωθεί δεν είναι αρκετά καλό. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε την συμφωνία η οποία τούτη τη στιγμή βρίσκεται υπό Είναι η νέα συμφωνία ενισχυμένη συνεργασίας με την Αστάνα και βεβαίως ε, και ε, η έκθεση για την στρατηγική ε, για την κεντρική Ασία που αφορά βεβαίως και το Καζακστάν ανεφέρετο ότι η ασφάλεια της περιοχής περνάει και την, από την ασφάλεια και τη σταθερότητα των πληθυσμών όπου φυσικά θα πρέπει να αναφερθούν τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν με ευχαριστεί καθόλου ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα. Κάποια στιγμή σίγουρα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιδράσει. Είχα την ευκαιρία να πω ότι όταν ένας ε, εκπρόσωπος αντιπολίτευσης όπως ο κύριος Κοσλόφ έρχεται εδώ και μιλάει ε, και μετά επιστρέφει στη χώρα του και τον ε, φυλακίζουν αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα και στα πλαίσια μιας άλλης συζητήσεως είχαμε πει ότι όταν μια χώρα είναι πλούσια, όπως το Καζακστάν, γιατί το Καζακστάν έχει μεγάλο πλούτο σε πρώτες ύλες, γι' αυτό ακριβώς θέλει εμπορικές σχέσεις ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θέλει επαφές με τη χώρα αυτή. Όταν μια χώρα λοιπόν είναι πλούσια θα πρέπει να έχει και πλούτο όσον αφορά την αντιμετώπιση ε, του πληθυσμού, όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις καζακικές αρχές. Έχουν κάθε δυνατότητα ε, να εφαρμόσουν ε, δημοκρατικές αρχές, να σεβαστούν τα συνδικάτα, να σεβαστούν τα μέσα ενημέρωσης, την ελευθεροτυπία κτλ. λοιπά. οι σφαγές που έλαβαν χώρα στην Κάναζάουζεν και ζητώ συγγνώμη γιατί το προφέρω άσχημα λέει η ομιλήτρια ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να ε, καταλάβουμε ότι είναι ε, πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή οι σφαγές και φυλακίσεις και βασανισμοί είναι απαράδεκτα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή συνάδελφε. Πολύ καλά τα είπατε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν οι σχέσεις, οι επικρίσεις μας ε, δεν αφορούν ε, προς εσάς, δεν αφορούν το γεγονός ότι ας πούμε δεν παρακολουθείτε ε, τις επιμέρους παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ότι η, ότι η ύπατη εκπρόσωπος αναφέρεται ε, στο ζήτημα μονάχα όταν μιλάει στο πανεπιστήμιο και σε φοιτητές αλλά θα πρέπει να κάνει και κάποιες δηλώσεις σε επίσημο επίπεδο. και πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μου διαρκώς γίνεται αυτή η συζήτηση. Δηλαδή λέμε ότι θα πρέπει να ε, αναφέρουμε σε χώρες πλούσιες όπως το Καζακστάν με τις οποίες θέλουμε ε, εμπορικές εταιρικέ σχέσεις θα πρέπει να αναφέρουμε πολύ συγκεκριμένα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα σας ξαναδώσω κυρία μου τα, τον λόγο αλλά για λίγο παρακαλώ. Ναι, ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ήθελα απλώς ε, να υπογραμμίσω ότι η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος ε, έχει αναφέρει το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και σε επίσημες δηλώσεις της. Και επίσης όσον αφορά την ετοιμιγορία κατά του κυρίου Κοσλόφ, επίσης η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος έχει κάνει συγκεκριμένη συγκεκριμένη δήλωση και μάλιστα εκπρόσωπος της ΕΑΣΕ είχε παρακολουθήσει την δίκη και η Λέδη Άστον έκανε συγκεκριμένη δήλωση ε, αναφέροντας ότι κατά την άποψή της αυτή η καταδίκη είχε πολιτικά κίνητρα. Ε, και πρέπει να σας πω ότι πέραν των όσων είπε στο Πανεπιστήμιο ε, όπου βρεθεί και όπου σταθεί και σε δημόσιο και σε ιδιωτικό χώρο και συζητήσεις αναφέρει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και με την ευκαιρία των δύο ε, ψηφισμάτων ε, και του 11 και του 12 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σχετικά με την συνεργασία με το Καζακστάν και όσον αφορά και τα συμπεράσματα της Επιτροπής Συνεργασίας τον Οκτώβριο του 2012 μας βρίσκουν σύμφωνους όλα αυτά τα, όλα αυτά τα κείμενα και επομένως βεβαίως θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η δημόσια συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε ε, στις 20 και 21 Φεβρουαρίου. Το επόμενο ζήτημα το οποίο αφορά ενημέρωση από τον ειδικό εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον διάλογο Αφρικανικής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν. Ευχαριστώ.